ήρθε η ώρα, και το επαναλαμβάνω αυτό, απευθυνόμενος προς τις χιλιάδες που θα διαδηλώνουν στην ε, Λισαβόνα να πούν ότι αρκετά πια. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις του ενός λεπτού και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έκθεση Ρίτα Μπορσελίνου σαν για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέσσερα λεπτά έχετε το λόγο κυρία εισηγήτρια. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, παρουσιάζω σήμερα την έκθεση πρωτοβουλία μου όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποια συγκίνηση. Αυτέ τι μέρε, με τα γεγονότα, έχουμε τα 20 χρόνια που σκότωσαν το δικαστή Φαλκόνε, την γυναίκα του και την συνοδεία του και όλα τα ήταν θύματα της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Και εκεί αφιερώνω την έγκριση αυτής της εκθέσεως και πιο συγκεκριμένα στην Μελίσσα Μπάση το νέο θύμα της απόπειρα που έγινε, του εγκληματικής ενέργειας που έγινε στον Μπρίντι, στο σχολείο του Μπρίντεζη το περασμένο Σάββατο και άλλες έξι κοπέλες τραυματίστηκαν. Δεν ξέρουν ποιο το έκανε, είναι άγνωστο, αλλά ε, δημιούργησε μια ένταση και ανασφάλεια ε, και τελικά και οργανισμοί και άτομα μπορούν να υποστούν βίες πράξεις. Και μερικές σκέψεις πάνε και στα θύματα της, του σεισμού στην Εμίλια Ρωμάνια, διότι ακόμα αφορά την εσωτερική ασφάλεια, ακόμα και φυσική καταστροφή. Το κείμενο που ψηφίσουμε αύριο υπογραμμίζει τη σημασία που έχει μια στρατηγική που είναι συνεκτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την σημαντική προσπάθεια που κατέβαλε στην επεξεργασία του κειμένου. Η ασφάλεια, όπως επανειλημμένα το τονίσαμε στην έκθεση, θα πρέπει πρέπει να την εγγυόμεθα ψευόμενη το κράτο δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι αναπόσπαστα τμήματα τη στρατηγική αυτή. Και γι' αυτό το λόγο έχει ιδιαίτερη σημασία ο ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που θα πρέπει να δραματίσουν σε αφορά τον καθορισμό και την εφαρμογή τη στρατηγική και συγκεκριμένα στο πλαίσιο που ακολουθεί τη Λισαβόνα, τη θήκη Λισαβόνα. Σε αυτό το πλαίσιο χρειάζεται να παίξει το ρόλο του τον απαραίτητο του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη φάση τη επεξεργασία των προτεραιοτήτων τη στρατηγική και στη φάση τη αξιολόγηση αυτών. Πρόκειται περί ρόλου που απορρέει από το ηθίες που έχει ένας νομοθέτης, πλήρης νομοθέτης που έχει όσον αφορά θέματα ασφάλεια στο Κοινοβούλιο και πρόκειται και βασικό στοιχείο για να εξασφαλίζει επαρκή έλεγχο δημοκρατικό που θα πρέπει να εφαρμόσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γι' αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να έχουμε τακτική επαφή μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Ένα κύκλο πολιτικό κοινοβουλευτικό που συνδέεται με την ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του ζητήματο και όπου καταλήγει σε μια ετήσια έκθεση του Κοινοβουλίου στον αφορά το πώ εφαρμόζεται η στρατηγική τη εσωτερική ασφάλεια. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει σαφή εικόνα όσον αφορά τι απειλέ για την εσωτερική ασφάλεια. Κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα. Θέλουμε η Ευρωπόλ μαζί με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και των διαφόρων φορέων να μπορεί να δραματίσει και να κάνει ανάλυση γενική των απειλών που πρέπει να αντιμετωπιστούν από την Ένωση μέσω μεθοδολογία πιο στέρεα και διαφανού με τη συνεισφορά πληροφοριών που θα δίνουν τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά του πέντε στόχου που έχουν προτεραιότητα και έχουν αναφερθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζουμε ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι εξαρτητικό ο κατάλληλο που παρουσιάζεται και πιθανότατα η σειρά των προτεραιοτήτων θα μπορούσε να έχει καλύτερη διάθρωση. Η καταπολέμηση τη τρομοκρατία, του οργανωμένου εγκλήματο και τη μαφία θα πρέπει να παραμείνουν για μα προτεραιότητε κλειδιά μια στρατηγική εσωτερική ασφαλεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω δεν θα πρέπει να ξέρει να αντιδρά, αλλά να ξέρει και να προλαμβάνει και θα πρέπει να προβλέπει και τι γίνεται στην Ευρώπη. Είδαμε τι έγινε στο Μπρίντεζι και αλλού. Θα πρέπει να μπορούμε να εντοπίζουμε σε έγκαιρη περίοδο τα σήματα ριζοσπαστικών πράξεων ε, και βαρβάρων πράξεων ε, του, ε, της βία. Η συνεργασία δικαστική είναι μεγάλη συνιστόσα τη αντική ασφάλεια. Περιγράφεται άλλωστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν. Κοινή δράση μεταξύ των δικαστικών αρχών ζωτική σημασία στην Ευρώπη για να αντισταθούμε στην τρομοκρατία και στην εγκληματικότητα και θα πρέπει να έχει προτεραιότητα. Είναι προτεραιότητα έχει καταπολέμηση της διαφθοράς, ε, το, το ε, έγκλημα κάτω περιβάλλοντος, ε, εγκλήματα οικονομικά και των επιχειρήσεων για να κατολεμήσουμε και την ε, εγκληματικότητα στο διαδίκτυο. Δεν δικαιολογείται ε, η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων που εισαγάγει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε Ασφάλεια. Ασφάλειας. Όπως είδαμε και με την άκτα, δεν είναι θέμα, είναι περίπλοκο θέμα που αφορά και τα δικαιώματα τα ατομικά και χρειάζεται μια ενδελεχέστερη συζήτηση. Λοιπόν, κλείνω ευχαριστώντα όλου και όλου εισηγητέ που συνέβαλαν στην σύνταξη αυτή τη εκθέσεω και θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω και τους υπαλλήλους των διαφόρων ε, πολιτικών ομάδων και την δική μου βοηθό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πάσκα, συνάδελφε Πάσκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν πολλές ε, απειλές για την εσωτερική ασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ε, εσωτερική ασφάλεια είναι η οργανωμένη εγκληματικότητα, το αναπτυγμένο οργανωμένο έγκλημα. πλήττεται το επίπεδο ζωής ε, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργείται το, η δυνατότητα για ε, παράνομο εμπόριο, για πορνεία, για εμπόριο ανθρώπων. Και γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε μία σύνθετη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εσωτερική ασφάλεια διαθρωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζουμε και την, ε, τις εξωτερικές σχέσεις και την εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό νομίζω ότι θα αποτελέσει βασικό πυλώνα για την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπασέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας ε, ανήκει σε ένα από τους ε, βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειάζονται και τα συγκεκριμένα μέτρα ώστε να επιτύχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους τους πολίτες, για κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχουμε πέντε βασικούς τομείς που έχουν επισημανθεί από την Επιτροπή, προτείνονται και συγκεκριμένα μέτρα και αποτελεί, αυτό αποτελεί ένα συγκεκριμένο θετικό βήμα. Χρειαζόμαστε όμως περαιτέρω προσπάθειες ε, για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και την εγκληματικότητα γενικότερα καταπολέμηση και μικρών μορφών ε, εγκληματικότητας όπως ε, μικροκλοπές ή κλοπές αυτοκινήτων. Πιστεύω ότι πρέπει να έχει ένα ισχυρότερο ρόλο η Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 6. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Και δίνω τώρα το λόγο στην Επίτροπο, την κυρία Μάλμστρομ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε καταδικάζουμε ε, και εμείς αυτά που έγιναν στον Πρίτεση το Σαββατοκύριακο. Uh, Ήταν πραγματικά αποτροπιαστικά όσα συνέβησαν και βέβαια η μετονομασία του σχολείου στο όνομα της ε, κυρίας ε, Φαλκόνε, της κοπέλας αυτής μάλλον, είναι κάτι το οποίο θα μας θυμίζει για πάντα αυτά τα γεγονότα. Ήταν βαρβαρότητα αυτό που συνέβη. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την έκθεσή σας, είναι εξαιρετική. Θέλω να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις και όλους τους βουλευτές ε, γιατί θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της στρατηγικής για την αστερική ασφάλεια που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι κοινή ατζέντη και για τα τρία θεσμικά όργανα και ο οργανισμός θα πρέπει να έχει σαφείς ε, αρμοδιότητες, καθήκοντα αλλά και κοινό στόχο γιατί η ασφάλεια των πολιτών είναι στο επίκεντρο όλων μα των προσπαθειών. Η στρατηγική εσωτερική ασφάλεια είναι η καλύτερη πλατφόρμα για την αντιμετώπιση απειλών ασφαλείας ένα σημαντικό σκέλος είναι και η επιχειρησιακή συνεργασία, κάτι που βλέπουμε και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Χαιρετίζουμε λοιπόν ε, αυτό τον κύκλο που θέλουμε να ε, θεσπιστεί, δηλαδή κοινό διάλογος με το Κοινοβούλιο, με τα Εθνικά Κοινοβούλια και με την εκπόνηση και την υποβολή τακτικών εκθέσεων από την Κομισιόν. Έχουμε τη δεύτερη έκθεση υλοποίηση, μέχρι τα τέλη του έτους θα δημοσιοποιηθεί. Η υλοποίηση τώρα τη ε, στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια ουσιαστικά έχει να κάνει με την ε, τήρηση των δεσμεύσεων που έχουμε να λάβει ε, σε πέντε τομεί για την καταπολέμηση και αποτροπή διεθνών εγκλημάτων, κυβερνοεγκλήματο, διαχείριση εξωτερικών συνόρων, αντιμετώπιση εθνικών καταστροφών κτλ. Είχαμε μία πρώτη δημοσίευση, είχαμε την έκθεση για την κατάσχεση αγαθών κάποια δίκτυα για την ευαισθητοποίηση σε σχέση με την ριζοσπαστικοποίηση και άλλες πρωτοβουλίες. Και θα έχουμε και μεταρρυθμίσεις για τη ΣΕΠΟΛ, την Europol και το Eurojust για να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ αστυνομικών υπηρεσιών και σε εθνικό επίπεδο Θέλουμε επίσης ε, να βελτιωθεί και η προστασία των κρίσιμων υποδομών. Μέχρι τα τέλη του έτους θα έχει διοργανωθεί και μια διάσκεψη στην οποία θα ανταλλάξουμε εμπειρίες ε, και θα αξιοποιήσουμε τα όσα έχουμε διδαχθεί όλον αυτό το χρόνο. Θα ακούσουμε ιδέες ε, για συγκεκριμένες πολιτικές. Στη δεύτερη έκθεση λοιπόν για την υλοποίηση θα δούμε τον απολογισμό της εκτέλεσης προηγούμενων δράσεων και θα εξετάσουμε δυνατότητες που μπορεί να μας προσφέρει η ασφάλεια για να ανταποκριθούμε και να αντιμετωπίσουμε και την οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αν θέλουμε να έχουμε ένα περιβάλλον όπου οι επενδυτές, ο κόσμος, οι εταιρείες να, να νιώθουν ασφαλείς. Η έκθεσή σας λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, λιθάρι σε αυτή την προσπάθεια για την επόμενη μιας στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας και θα συνεργαστούμε μαζί σας με πολύ μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπε. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση επί του θέματος αυτού. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε τώρα την έκθεση Κορνέλης Δε Γιόγκ όσον αφορά την προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όσον αφορά